Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη που αφορά την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο με θέμα δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα. Είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που έχει υποβάλει το προφορικό ερώτημα και θα ήθελα να καλωσορίσω την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Παναγιώτοβα, και να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέγνερ, τη συντάκτρια της ερώτησης αυτής. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρία Παναγιώτοβα, στις 4 Ιουλίου 2017 το Κοινοβούλιο εξέδωσε την απόφασή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δημόσια υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ο δημόσιος έλεγχος της φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και η πρόθεση εταιρικής ευθύνης με την επιβολή απαιτήσεων γνωστοποίηση σε ορισμένες εταιρείες. Η ισχυρή σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις εταιρικές εκθέσεις οδήγησε την Επιτροπή να επιλέξει τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας. Με νομική βάση το άρθρο 50 παράγραφος 1. Η απόφαση του Κοινοβουλίου, βασισμένη στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Τη 12 η Ιανουαρίου 2017 συμφωνεί με την επιλογή τη Επιτροπή για την νομική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι μιλάμε εδώ πέρα για ζητήματα διαφάνεια, για ζητήματα νομική βάση και κυρίω για χρηματοπιστωτικέ διατάξει. Με άλλα λόγια μιλάμε για του λογαριασμού των εταιριών και δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για ένα νέο φόρο εισοδήματο. Πρέπει λοιπόν εμεί να διαπραγματευτούμε μαζί σας με το Συμβούλιο. Εμείς είχαμε θελήσει να ολοκληρώσουμε διαδικασία μέχρι πέρυσι, αλλά εσεί στο Συμβούλιο δεν προχωρήσατε ακόμα καθόλου. Ορισμένοι Υπουργοί Οικονομικών θεωρούν ότι πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την φορολογία και ότι θα πρέπει να ισχύει το άρθρο 115 της συνθήκης. Είναι σαφές ότι στόχος δεν είναι η ενοποίηση των ε, φορολογικών συντελεστών, αλλά η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών. Στόχος είναι να υποχρεωθούν οι μεγάλες εταιρείες του πλανήτη να υποβάλουν ανοιχτά και δημόσια στοιχεία για τη φορολογική τους τακτική. Αυτό ε, αποτελεί και τον πυρήνα του, του κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να δεσμεύει όλες τις πολυτεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούν στην Ευρώπη. Έλεγχος από, την, από τις δημόσιες αρχές, τις κρατικές αρχές. Πώς αιτιολογεί το Συμβούλιο βάσει των ε, ε, διεθνών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι ε, έχουμε υιοθετήσει ηγετικό ρόλο στο Financial CBCR. Και παραπέμπω εδώ και στον σχετικό, στη σχετική οδηγία. Θέλετε να ακολουθήσετε ένα σύστημα Τραμπ. Πώς αιτιολογείτε τις διετής καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί. Πώς αιτιολογείτε τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την νομική βάση. Είναι σαφές στους υπουργούς ότι δεν μιλούμε για απλώς για τα ποσά που θα καταβάλουν ως ε, φορολογία οι μεγάλες εταιρείες αλλά τους κανόνες. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε εντός της τρέχουσας θητείας να σημειώσουμε πρόοδο. Φυσικά και πρέπει να δεσμεύονται και να υποχρεούνται σε διαφάνεια οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται. Μόνο για τις μεγάλες μιλούμε. Για, ε, για εκείνες που κάνουν κύκλο εργασιών πάνω από 57 εκατομμύρια ε, ευρώ. Νομίζω ότι από πολλές απόψεις η συζήτηση αυτή είναι απλά προσχηματική ε, προκειμένου να ροκανιστεί ο χρόνος, να ξεχαστεί η υπόθεση. Ρωτήστε τις Ρωτήστε τους ε, αυστριακούς συναδέλφους σας γιατί μπλοκάρουν αυτό το νομοθέτημα. Τόσο πολύ αγγίζει το, η νομική αυτή πράξη τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Δεν, προστατεύεστε, ε, δεν, δεν ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε τις μεγάλες, ούτε τις startup προστατεύεται μόνο τους κολοσσούς που μέχρι τούδε δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους. Και αυτό είναι αδικία απέναντι στους ε, φορολογούμενους πολίτες της Ευρώπης. Και έχουν δικαίωμα οι φορολογούμενοι της Ευρώπης να γνωρίζουν πόσους φόρους πληρώνουν στην Ευρώπη το Facebook, η Starbucks, η Amazon. Και γι' αυτό θέλω να σας καλέσω στο Συμβούλιο να αναλάβετε επιγόντως δράση. Ε, Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η Υπουργός, κυρία Παναγιώτοβα, που εκπροσωπεί το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέγνερ ε, και τον κύριο Σφόμποντα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιούρη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και η Κομισιόν έχει υποβάλει από το 2016 μία ε, πρόταση για να αποφύγουμε τη διάβρωση φορολογικής βάσης. Το Συμβούλιο εξέτασε σε πάνω 50 συνεδριάσεις του, συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και υπό την σκέπη τεσσάρων διαδοχικών προ... Προ... προεδριών αυτό το θέμα. Ο κ. Γκουαλτιέρ και ο κ. Βόμποντα έγραψαν επιστολή στον πρέσβη μας ε, ρωτώντα που βρίσκεται το θέμα και ζητώντας να επιταχυνθούν οι εργασίες. Απαντήσαμε σε αυτή την επιστολή, πενθυμίζοντας ότι υφίστανται ανεπίλητα πολιτικά θέματα τα οποία δυσκολεύουν συμφωνία στο Συμβούλιο. Ένα από αυτά είναι η φορολογική βάση που προτείνεται. Αυτό το ζήτημα αμφισβητεί ακόμα και την εφαρμογή της ε, τακτικής διαδικασίας ε, νομοθεσίας. Ε, συνεχίζουμε τις ε, τεχνικές εργασίες που ήταν ήδη αρκετά προχωρημένες από τις προηγούμενες προεδρίες και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις με τις αντιπροσωπείες για να ξεσκαλώσουμε το φάκελο αυτό. Καταλαβαίνετε όμως, όμως ότι δεν μπορώ να αναλάβω κάποια συγκεκριμένη δέσμευση σήμερα. Το Συμβούλιο νομίζω ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διευκρινίσει τη θέση του. Θα σας ενημερώνω για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Να σας βεβαιώσω ότι εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ποσπίσιλ έχει το ρολόγιο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου και πραγματικά σοκάρει η απάντησή σας. Δεν υπάρχει καθόλου και την απορρίπτω. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται εδώ πέρα μία πρόφαση, ένα άλοθη, για να μην πείτε ουσιαστικά τίποτα. Έχουμε μία πρόταση οδηγίας, αυτή θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Είναι για το κοινό συμφέρον αυτό. Το είπατε κι εσείς η ίδια, ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και στο Συμβούλιο κάντε το παν για να μην εγκριθεί αυτή η πρόταση οδηγίας χρησιμοποιείτε δήθεν ένα επιχείρημα για νομική βάση με την οποία δεν συμφωνείτε, μα τι δικαιολογία πραγματικά είναι αυτή ουσιαστικά θέλετε να μπλοκάρετε την όλη διαδικασία. Θα ήταν πολύ πιο ειλικρινέ να λέγατε ότι υπάρχουν χώρε στο Συμβούλιο οι οποίε δεν θέλουν να εγκρίνουν αυτή την πρόταση οδηγία. Να βγουν λοιπόν δημόσια έξω και να μα πούνε ότι δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση οδηγία και ουσιαστικά δεν θέλουν να γνωστοποιήσουν περαιτέρω πληροφορίε για τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του. Και τότε πραγματικά οι πολίτε θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ στους ψηφοφόρους μου να εξηγήσω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαμάχη για την νομική βάση και για ποιο λόγο τόσο σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αυτή τη στιγμή δεν γνωστοποιούνται επειδή δεν το επιθυμούν ουσιαστικά ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει οι χώρε αυτέ να βγούνε και να το πούνε ξεκάθαρα αυτό προ τα έξω, χωρί να κρύβονται πίσω από δικαιολογίε. Ο κύριο Κοφεράτη έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Κυρία Υπουργέ, το είπατε και εσείς ίδια, έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας ζητά να εγκριθεί αυτή η πρόταση οδηγία που συζητήσαμε και εγκρίναμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή την δυνατότητα υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τι μεγάλε πολυεθνικέ επιχειρήσει. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε περαιτέρω την απόφαση αυτή. Επίση, τα τελευταία αυτά χρόνια είδαμε τόσα πολλά σκάνδαλα, τα οποία καταδεικνύουν ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιοφυγή αποτελούν τεράστιο φαινόμενο που επηρεάζει πραγματικά πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα και την κατανομή πλούτου σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολυεθνικέ αυτέ επιχειρήσει κάνουν τεράστια κέρδη, πληρώντα ελάχιστου φόρου. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια οδηγία που να επιβάλλει στι επιχειρήσει αυτέ την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων όσον αφορά το φορολογικό του εισόδημα. Χωρί τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν αυτές οι απαράδεκτες, άδικες συνθήκες για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες είναι νομοταγείς και οι οποίες καταβάλουν τους φόρους τους. Περιμένουμε λοιπόν πολύ γρήγορα μια θετική ανταπόκριση από το Συμβούλιο στο έτοιμά μα αυτό. Πραγματικά νιώθω ντροπή, κυρία Υπουργέ, ως Ευρωπαίος νομοθέτης. Βρισκόμαστε ενώπιον μια συγκεκριμένη κατάσταση που τη γνωρίζετε. Είναι μια δραματικότατη κατάσταση. Έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν το φόρο τους και να σέβονται τους κανόνες. Και από την άλλη μεριά έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις που κρύβονται πίσω από μια θολούρα και καταφέρουν και φοροδιαφεύγουν. Το ζητούμε εδώ και δύο σχεδόν χρόνια μετά από διαβουλεύσεις με τους πολίτες, μετά από σκάνδαλα που έγιναν. Ζητούμε με τη στήριξη των δύο νομικών υπηρεσιών, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου, να προχωρήσουμε προς μια δημοσιοποίηση πληροφοριών, μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι θέμα πληροφόρησης, δεν είναι θέμα φορολογίας. Μην κρύβεστε πίσω από αυτό το τεχνικό επιχείρημα για να μην δράσετε. Παρακαλώ πολύ, πάρτε το θέμα στα χέρια σας. Thank you. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε σε τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη φορολόγηση των πολυεθνικών ιδίως εταιριών. υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες οι οποίες αλλού παράγουν αλλού πολλούν τα προϊόντα τους με μεγάλα κέρδη και αλλού φορολογούνται με εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές. η επιβολή υποχρέωσης για δημοσίευση δηλώσεων των πολυεθνικών εταιριών με πληροφορίες ανά μπορεί να προάγει την εταιρική ευθύνη και να περιορίσει τη αποφυγή μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε βιώσιμο να επιβαρύνονται με ολοένα και πιο δυσβάστακτους φόρους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ενώ να απαλλάσσονται κατ' ουσία οι μεγάλες πολυεθνικές. κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό είναι αδικαιολόγητη. Για 1,5 λεπτό, κύριε Ροζάτη. Ευχαριστώ πολύ. Η φορολογική διαφάνεια αποτελεί κρίσιμη σημασία ζήτημα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα, Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα πριν από δύο χρόνια το 2016. Εγώ ήμουν σκιώδης του ΕΛΚ για αυτή την υπόθεση και έπειτα από μήνες σκληρής δουλειάς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα την διαφάνεια και την προστασία των επιχειρήσεων. Εγκρίναμε την απόφασή μας πέρσι τον Ιούνιο. Τώρα ε, κηρύσσοντας την ε, δέσμευσή μας στην, και παρά την, το γεγονός ότι κηρύσσει τη δέσμευσή της ε, στη φορολογική διαφάνεια η Προεδρία δεν έχει κάνει τίποτα. Το να μπλοκάρεται αυτός ο φάκελος γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αποφασίσουν επί της νομικής βάσης δεν είναι σοβαρή τακτική. Εδώ δεν μιλάμε για οδηγία για φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικά ποσά που θα καταβάλλονται. Μιλούμε απλώς για ε, κανόνες. Ε, δεν περιορίζονται οι εθνικές αρμοδιότητες. Γι' αυτό και καλό το Συμβούλιο να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προχωρήσει η διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό η κυρία Σλάιν. Δέκα μήνες πέρασαν από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας για την δημόσια υποβολή εκθέσεων αναχώρα ένα πολύ σημαντικό θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ένα εργαλείο διαφάνειας με μικρό κόστος, το οποίο θα πετούσε από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Που θα πετούσε από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως άλλωστε προβλέπεται από, για το τραπεζικό τομέα από την κοινοτική νομοθεσία, να δημοσιοποιούν για κάθε υποκατάστημά τους σε κάθε χώρα στοιχεία όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ακόμα περιμένει να συνεργαστεί με εσά στο Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει από εσά σε μια κοινή θέση. Αυτή τη στιγμή τα όσα μας λέτε για νομική βάση αποτελούν απλώς μια δικαιολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε να προχωρήσετε σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. LuxLeaks, Paradise Papers, Panama Papers, πόσα σκάνδαλα ακόμα πρέπει να δούμε για να δούμε ανταπόκριση από το Συμβούλιο. Διακόπτη, Πρόεδρο. Σα ζητώ συγγνώμη, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, λέει Πρόεδρο στην Ευρωβουλευτή. Ολοκληρώστε το λόγο σα. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ αλλά γενικά μιλάτε λίγο πιο αργά ώστε να μπορούμε να σας παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη δικασία Κάτσθια. Έχουμε δύο, μιλητές. δύο μιλητές. κυρία Πιετικά είναι πρώτη. Παρακαλώ. Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία νομικών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί κοινής αρμοδιότητας όσον αφορά τους λογίστε ε, τους λογιστικούς ελέγχους και τις σχετικές οδηγίες. Το να ισχυρίζεται λοιπόν κανείς ότι θα υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένης νομικής βάσης είναι ένα φύλλος που προσχηματικά και σκόπιμα χρησιμοποιείται προκειμένου να μπλοκαριστεί αυτή η ε, πλέον ανάγκη να υποβάλλονται εκθέσεις αναχώρα. Αυτό αντίκειται σε κάθε αίσθημα δικαίου που αισθάνονται οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Ελπίζω πραγματικά η Βουλγαρική Προεδρία να συγκαλέσει συνεδρίαση και να ζητήσει την νομική γνωμοδότηση διαφόρων φορέων ε, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το ζήτημα στο Συμβούλιο, διότι το να καθόμαστε και να το κοιτάμε το θέμα αυτό δεν, ε, δεν πρόκειται να μας φέρει σε λύση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την ώρα που οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους και μάλιστα έχουμε σε πολλές χώρες όπως την Ελλάδα μια τεράστια φορομπηκτική πολιτική, οι πολυεθνικές φόρο και φόρο αποφεύγουν το παράδειγμα με τα luxleaks είναι καθοριστικό. τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; πρέπει οι πολυεθνικές να φορολογούνται εκεί που βγάζουν τα κέρδη και φυσικά η οδηγία η οποία θα υποχρεώνει να υπάρχει δημοσίευση εκθέσεων για τα κέρδη κάθε πολυεθνικής για κάθε χώρα νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στο χτύπημα της φοροδιαφυγής. δυστυχώς συγκεκριμένα κράτη όπως είπε και η βουλγαρική προεδρία έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία και σας ρωτώ κυρία παναγιώτοβα ποια κράτη μέλη έχουν μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία να τα ονομάσετε. και σας ρωτώ η ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στα κράτη μέλη που έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία έγκρισης της οδηγίας. θέλουμε διαφάνεια θέλουμε απαντήσεις εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στην κυρία Παναγιώτοβα για να απαντήσει. Παρακαλώ. I think it's working. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακολούθησα προσεκτικά και σημείωσα όλες τις παρατηρήσεις σας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας ε, στο φάκελο αυτό. Εγώ εδώ εκπροσωπώ όλα τα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου δεν μπορώ να κατονομάσω συγκεκριμένες χώρες και τη στάση τους. Το πρόβλημα δεν είναι η διάσταση απόψεων στο Συμβούλιο. Αυτό που χρειάζεται πάντοτε είναι ε, χρόνος για να ε, εξασφαλίζεται συμφωνία και στις Βρυξέλλες αλλά και στις ε, εθνικές πρωτεύουσες προκειμένου να οριστικοποιήσουν οι χώρες τη θέση τους. Ξέρετε ότι χρειαζόμαστε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Η Βουλγαρική Προεδρία ε, προτίθεται να καταβάλει προσπάθειες ώστε να προχωρήσει το θέμα, να σημειωθεί πρόοδος και όπως είπα και εισηγητικά, εμείς ε, είμαστε ανοιχτοί για περαιτέρω συζητήσεις στο θέμα αυτό και όταν σημειωθεί πλέον πρόοδος ε, θα διοργανώσουμε και μια σχετική συνεδρίαση μαζί σας. Προσωπικά όμως σας διαβεβαιώ ότι είμαι στη διάθεσή σας και για διμερείς επαφές αν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.